απέτυχε το σύστημα Spitzenkandidat. Ο κύριος Ντέμπερ κάθεται εκεί πίσω, ενώ θα έπρεπε να κάθεται μπροστά. Μικρό βήμα για σας, αλλά μεγάλο το άλμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατ' ουσίαν, αυτά που ακούσαμε σήμερα ήταν η κηδεία του συστήματος Spitzenkandidat και βρισκόμαστε στο δρόμο των ε, ματαιωμένων ε, ονείρων. Άκουσα, κάνατε υποσχέσεις ε, προς όλους ε, και προς τους πράσινους. Κατ' ουσίαν, περί τίνος πρόκειται. Λέτε ότι όλα αυτά είναι αξίες, οι οποίες πρέπει όμως αξίες να εφαρμοστούν στην πράξη. Όσον αφορά το στρατό. Εκεί υπήρξαν, ε, το γερμανικό αναφέρομαι, αλλά υπήρξαν ε, κάποιες ε, τυχείς εξελίξεις, αλλά και εσείς ευθέτε για αυτά που συνέβησαν. Αν κάτι δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε και εκεί θα αποδώσετε την ευθύνη σε άλλους. Εγώ θα έλεγα το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη. Ένα λεπτό ο κύριος ε, Βίλιομσεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ε, θα ψηφίσουμε κατ' ουσίαν για το κλίμα. Βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ οξία κλιματική κρίση και αυτό που διακυβεύεται είναι κατά πόσον θέλουμε να έχουμε μια πολιτική άμβλυνση του προβλήματος ή όχι. Ακούσαμε την απάντηση από τον κυρία Φοντελάιν σήμερα, η απάντηση ήταν ένα ξεκάθαρο όχι. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα όχι, 50% μείωση των ε, εκπομπών του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Δεν αρκεί αυτό για να αποφύγουμε κλιματική καταστροφή. Ούτε και το 55% αρκεί για να αποφευχθεί αυτή η καταστροφή. Την ε, κλιματική δράση την χρειαζόμαστε αμελητή και γι' αυτό το λόγο εγώ θα καταψηφίσω την κυρία Πόντερ Λάιν και καλώ όλους εσάς που είστε υπέρ της κλιματικής αλλαγής να κάνετε το ίδιο. Έχει έρθει η στιγμή, αν σήμερα ψηφίσετε όχι, αυτό θα σημαίνει δράση. Δράση που θα συνοδεύουν τα λόγια μας. Ψηφίστε για το κλίμα, ψηφίστε για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής, καταψηφίστε την κυρία Ποντελάν σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιντσίτς, για 1,5 λεπτό. Κυρία Φοντελάιν, πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβιώσει την επόμενη οικονομική κρίση. Εσεί αντιπροσωπεύετε όλα όσα πάνε στραβά στην Ευρώπη. Την ε, κεντρικοποίηση, το έλλειμμα το δημοκρατικό, την οικονομική ηγεμονία. Εδώ μιλάμε για κεντρικοποίηση και συγκέντρωση. Πριν από κάποιο καιρό η Ιταλία ε, τον Εύδο πρόεδρο, ε, Ιταλό πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, ενώ 15 περιφερικές χώρες συμπεριλαμβανόμενες της Κροατίας δεν είχαν κανένα. Η κατάσταση είναι ίδια και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Πότε θα έρθει η σειρά κάποιου άλλου, της Μάλτας, της Κροατίας, της Σλοβακίας. Ποτέ όταν πρόκειται για τη δημοκρατία έρχεστε εδώ, στέκεστε ενώπιόν μας και δεν, έχετε, δεν έχετε νομιμότητα. Ποια εκλογική διαδικασία, ε, σε ποια εκλογική διαδικασία συμμετείχατε, πώς μπορείτε να έχετε νομιμότητα, πώς μπορείτε να ζητήσετε από τόσους ψηφοφόρους την νομιμότητά σας. Εδώ η διαδικασία δεν είναι δημοκρατική, συμφωνήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες και όλες οι ισχυρές δυνάμεις αποφάσισαν. Οι Γάλλοι θα πάρουν την κεντρική τράπεζα, οι Βέλγοι το Συμβούλιο και τίποτα για την περιφέρεια. Εσείς μιλάτε για τη Συρία, ότι πήγατε στη Συρία ή ότι δεχτήκατε το φιλοξενήσατε ένα παιδί από τη Συρία. Μπράβο σε εσά, αλλά από την άλλη πλευρά μιλάτε και για το ΝΑΤΟ ε, που συνεχώς προκαλεί αστάθεια και τις υπερηλαστικές δυνάμεις που δεν εξυπηρετούν την ειρήνη. Η Κροατία δεν έχει κανένα όφελος από αυτά. Ε, θα πρέπει να είστε ειλικρινείς, αλλιώς δεν θα πάρετε τη ψήφο, μου. Δύο λεπτά ο κύριος Μπελαμή. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Βαντελάγιο, ο Σεφ έλεγε ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος ε, να ε, βλέπουμε πραγματικά αυτό που βλέπουμε, να έχουμε το θάρρος και να βλέπουμε την κατάσταση ω έχει. Έχουμε απέναντί μας πολλές προκλήσεις, μετανάστευση, εμπορικές συμφωνίες κλπ. Ο πολιτισμός μας ο ίδιος παίζεται σήμερα και δεν είναι δυνατόν να δώσουμε καμία καμία οδό διαφυγής ε, στον εθνικισμό και τον λαϊκισμό. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Να μην υποβληθούμε πλέον σε ε, ε, στην παγκοσμιοποίηση και τις χειρότερες επιπτώσεις της. Λυπούμε σχετικά με τους γεωργούς. Δεν έγινε λόγο σήμερα το πρωί στην Γεωργία που είναι η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποτέ εμείς εδώ στο ΕΛΚ δεν θα δεχτούμε να γίνει απλώς ένα στοιχείο ε, στην εξίσωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, μεγάλες προκλήσεις. Ε, υπόθηκε και σήμερα το πρωί η Ευρώπη θα πρέπει να ε, εφαρμόσει έναν φόρο διοξιδίου του άνθρακος για τις χώρες που εξάγουν. Η Ευρώπη επίσης αντιμετωπίζει την μεταναστευτική κρίση. Ναι, κάθε θάνατο στη Μεσόγειο είναι τραγωδία. Αλλά ναι και κάθε τραγωδία αυτή είναι αποτέλεσμα της δικής μας διστακτικής στάσης. Ε, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Ευρώπη γιατί ε, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να φτάσουν παράνομα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε ε, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποδοχή, το, το, να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους αυτούς δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υφιστάμεθα τα πάντα. Εμείς έχουμε μια θαυμάσια Ευρώπη Κυρία Φόντερ Λέγεν, πρέπει να σώσουμε το μέλλον της. Ε, αυτό το μέλλον παίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα επόμενα πέντε χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ζητήσω τα επόμενα πέντε χρόνια να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Πύρη για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, κυρία Φόντερ Λέγεν η προσέλευση στις ευρωεκλογές ήταν η ψηλότερη που είχαμε στις κάτω χώρες. Είχαμε μια έντονη εκστρατεία, προσπαθήσαμε να πείσουμε ε, τους ψηφοφόρους και στο τέλος οι ψήφοι ήταν ε, αισιόδοξοι. Αλλά ε, και για το πώς θα πειράσουν την, τον νέο ε, επικεφαλής της Επιτροπής. Είχαμε μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτή η μεγάλη πλειοψηφία θα ε, υποστήριζε μόνο έναν από τους πίτσεν καντιντάτεν για την θέση της Επιτροπής. Ε, μετά όμως ξεκίνησε μια τόμπολα και η βγήκε το δικό σας όνομα από, ε, χωρίς να το περιμένουμε. Υπάρχουν φήμες για τις κάτω και νιώθει ο κόσμος ότι εξαπατήθηκε. Λένε γιατί ψηφίσαμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό στο Συμβούλιο διαδικασία του Spitzen ε, Candidate ε, καταπνίγηκε από τον Βίκτορ Ορμπάν. Ε, οι Πολωνοί, νέες, οι κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας είδαν την υποψηφιότητά σας ως νίκη. Εσείς δεν φταίτε γι' αυτό, αλλά το γεγονός ότι το είπαν το καθιστούν πιο σημαντικό ότι υιοθετείτε ξεκάθαρη θέση για το θέμα του κράτους δικαίου. Άρα η ερώτηση είναι, στηρίζεται τις διαδικασίες του άρθρου 7, όπου πρόσφατα η Επιτροπή και το Συμβούλιο ξεκίνησαν ενάντια ε, στις κυβερνήσεις Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Είναι σημαντικό να να, εκφράσετε τις αμφιβολίες και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αν θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο δημοκρατική. Θα απαιτηθούν τεράστιες προσπάθειες από πλευρά σα και από δικιά μας πλευρά. Κύριε Φοντενάιαν, στην ομιλία σας ε, παραθέσατε σημεία τα οποία ε, προσελκύουν τους προοδευτικούς ψηφοφόρου. Αν εκλεγείτε σήμερα, πιστεύω ότι μπορείτε να ε, βασιστείτε στη στήριξη του Ολλανδικού κόμματος σε ό,τι αφορά την πιο και η Ευρώπη. Κύριε ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρία Φοντερ Λάγεν πολλά υπόθηκαν ήδη για την μετανάστευση, το κλίμα, το κράτος δικαίου. Γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Είναι γεγονός ότι ε, όλα τα στοιχεία αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας ε, και ε, θα πρέπει εσείς να ξανασυνδεθείτε με το Κοινοβούλιο και μετά με τους πολίτες. Δεν είστε υπεύθυνοι, κυρία Φοντερλάγεν, αλλά θα πρέπει να θυμίζουμε αυτό το προπατορικό αμάρτημα το πούμε έτσι, ε, γιατί είχαμε ένα είδος μερκάτο και αυτό αποτέλεσε πραγματικά μια μεγάλη πληγή ε, και νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να κλείσουν οι πληγές με την μελλοντική διαβούλευση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, ψήφι ψηφιοποίηση, ρομποτική, ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, προωθήσουμε όλα τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε η Ευρώπη να βρει ηγετική θέση. Υπάρχουν συγχωνεύσεις οι οποίες δεν προχώρησαν καλά και που ακόμα μας πονούν πολύ. Η υγεία, δεν το γνωρίζετε εσείς κυρία Φοντερ η υγεία ε, ήταν πραγματικά ο φτωχός συγγενής ε, της προηγούμενης ε, Κομισιόν. Όσον αφορά τις σπάνιες αρρώστιες, δεν προωθήθηκε καθόλου το θέμα. Το, η διασυνοριακή αντιμετώπιση της υγείας. Πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε και για αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χαουτάλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φοντερ Λάιν, Είμαι ευτυχής ε, που αναφέρεται στις ε, πολιτικές ε, κατευθυντικές γραμμές ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός. Ο στόχος είναι να προσφέρει ευημερία στην ε, χώρα που ασχολείται με εμπορικές ανταλλαγές, αλλά όλοι γνωρίζετε ότι με εισαγωγή προϊόντων εξάγουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάμε για σκλαβιά, για αποψήλωση των δασών. Εσείς λοιπόν θα στηρίζατε υποχρεωτική ευρωπαϊκή νομοθεσία για ε, ολιγορία εκ μέρου ε, των επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μία δεύτερη ερώτηση. Εγώ έρχομαι από την Βόρεια Ευρώπη και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κλιματική αλλαγή έχει ολέθριες συνέπειες ε, στην Αρκτική. Η δική σας σε διάταξη για την Ευρώπη δεν αναφέρεται καν στην Αρκτική. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ερωτώ την πολιτική για την Αρκτική θα τη θεωρήσετε ως προτεραιότητα για τη νέα ε, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπέρκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, ως νεοεκλογής ε, Ευρωβουλευτής. Ε, μέχρι τώρα πρέπει να σας πω, εξεπλάγει από όλη αυτή η διαδικασία που επελέγει για τον σπίτσαν καντιντάτ. Και είναι λυπηρό το ότι πολλοί πολίτες της Ευρώπης αγνοήθηκαν και το μόνο που παίζει ρόλο είναι ότι λαμβάνονται αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Αυτό δεν, εμφυσί, δεν εμφυσά εμπιστοσύνη, αλλά προκαλεί αγανάκτηση. Και οι επιφυλάξεις μου αφορούν την εσωτερική ασφάλεια, τον έλεγχο των συνόρων, αφορούν κυρίως ε, την απειλή από την διεθνή μουσουλμανική ε, τρομοκρατία Είδαμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα από την πολιτική των ανοιχτών θυρών στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είδαμε το τι σημαίνουν αυτά για το προσωπικό, για την αστυνομία που και αυτή υποφέρει από τις περικοπές. Επειδή λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει ανεξέλεγκτη μετανάστευση και αυξάνεται ο κίνδυνος για επιθέσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα προβλήματα της ασφάλειας αντί να γίνονται λιγότερα, γίνονται περισσότερα. Κύριε Φοντελάν, θέλω να πιστεύω ότι όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, αυτά που είπατε δεν ήταν κενά λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κανκό, για ένα λεπτό παρακαλώ. Καλημέρα σας, ε, κυρία Φοντελάιν, Λέγομαι Ισίτα Κάνκο και είμαι ένα από τα επτά παιδιά μιας γυναίκας που αναγκάστηκε να φύγει όταν αποφάσισε να ε, ζητήσει διαζύγιο. Όταν γεννήθηκε η τελευταία μου αδελφή, η μητέρα μου ήταν 37, εγώ γίνα 39 και έχω μόνο ένα παιδί, δική μου επιλογή βέβαια, αλλά ξέρετε γιατί, διότι το να γεννήσει μια γυναίκα με ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ είμαι μια τέτοια γυναίκα. Είμαι φλαμαντή. Είμαι γυναίκα. Ε, όταν ήμουνα μικρή δεν ε, έφυγα ανησυχώ ως μητέρα στην Ευρώπη κλείνουμε τα μάτια όταν ο μουσουλμανισμός αρπάζει τις γυναίκες αγνοούμε την Μουράτ και άλλες γυναίκες αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλές εκείνες οι οποίες είναι αναγκασμένες να εφίσταται τις συνέπειες στην Ευρώπη. Βλέπουμε τι γίνεται με τον, Ισλαμικό ε, ριζοσπαστισμό. Πού είναι λοιπόν οι αξίες μας και εσείς ε, πώς θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη θέση σας για να προστατέψετε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα με τη θρησκεία τους. Το άρθρο 1 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται ακόμα σε αυτές τις γυναίκες. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε σε μια ισχυρή Ευρώπη, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ τους ανθρώπους και μην ξεχνάτε εκείνους που αποδίδουν αξία και σεβασμό στην επικουρικότητα. για ένα Κυρία Βαντερλάγεν, τι θα πείτε σε αυτά τα εκατομμύρια, πάνω από 100 ε, των ε, πολιτών που δεν σας ψήφισαν. Ποια θα είναι η νομοποίησή σας ε, για να αντιμετωπίσετε την κλιματική κρίση και την κλίση των ανισοτήτων. Θα μας πείτε ότι τα ταμεία είναι άδεια όπως η προκάτοχή σας ότι δεν υπάρχουν χρήματα ε, ενώ για άλλες πολιτικές υπάρχουν ε, γιατί βρίσκονται τα χρήματα αυτά εις ε, τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι το, η επιταγή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στέλνει στην Google, στην Amazon, ε, που στέλνονται στη, στους παραδείσους, στους ε, φορολογικούς. Όπως έλεγε ο Βίκτορα Σουγκό, ε, ο, η κόλαση των φτωχών κάνει το παράδεισο των πλουσίων και σε αυτό το παράδεισο βρίσκεται η νέα πρόταση, πρόεδρος. Εσείς κυρία Φόντερ Λέγεν. Ε, δεν θα, θα, αναλάβετε δράση κατά των φορολογικών παραδείσων όπως η Μάλτα ή το Λουξεμβούργο. Είστε η δική τους υποψηφία κυρία Φόντερ Λέγεν. Δεν είσαστε η υποψήφια των ευρωπαϊκών λαών. Κανένας ε, ε, ε φτωχός δεν σας πιστεύει. Εσείς είστε η, η, εικόνα των, του, της κόλασης των φτωχών. Εμείς αυτή την επιταγή προτιμούμε να τη σκίσουμε χαρά να σας ψηφίσουμε. For and a half minutes, Mr. Ενάμιση λεπτό ο κύριος Νικόλαος ε, Αλαβάνο. Ο κύριος Αλαβάνος. Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού στο πλαίσιο των ανταγωνισμών που οξύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της χαμηλής απόδοσης που καταγράφει η ευρωπαϊκή οικονομία. Ανεξάρτητα από αντιπαραθέσεις, όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος η νέα κομισιόν θα συνεχίσει τη βασική στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης ενίσχυση της κερδοφορίας των μονοπωλίων περιορισμός λαϊκών ελευθεριών φακέλωμα αντικομουνισμός τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη στρατιωτικοποίηση υπεριαλιστική επιθετικότητα που ενισχύει επικίνδυνους σχεδιασμούς και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Τουρκία στο αιγαίο στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. μετά ακριβώς την ανάδειξη της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση της χώρα μας το eurogroup συζήτησε την πορεία της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια των συμφωνηθέντων με την κυβέρνηση σύριζα με φόντο την τέταρτη αξιολόγηση και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. 2023. κομισιόν και eurogroup εντοπίζουν σειρά δημοσιονομικών κενών απαιτούν απαρέγκλητη τήρηση του 3,5% των πρωτογενών πλεονασμάτων των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας δηλαδή νέα βαριά μέτρα στις πλάτες του ελληνικού λαού κόστους 4,5 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν βάση για την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προβλέπουν γενίκευση πληστηριασμού λαϊκής κατοικίας, αύξηση φοροεισπρακτικών μέτρων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, νέες περικοπές στις συντάξεις, σε επιδόματα, ιδιωτικοποιήσεις, μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση υγείας πρόνοιας και εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι σε Ελλάδα και Ευρώπη πρέπει να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα, να οργανωθούν, να διεκδικήσουν τα σύγχρονα δικαιώματά τους στη δουλειά στη ζωή στη μόρφωση των παιδιών τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εσείς αναφερθήκατε σε μια πολιτική για το μέλλον της Ευρώπης ε, που σε μεγάλο βαθμό την ε, στηρίζουμε. Πρέπει να έχουμε μια τέτοια πολιτική οικονομική, οικονομική πολιτική που να βασίζεται στην πραγματική οικονομία. Χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική που θα έχει ως στόχο όπως και στην περιβαλλοντική πολιτική το 20% του ΑΕΠ να προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τη γεωργία. Όταν λοιπόν θα είσαστε πρόεδρος της Επιτροπής να εφαρμόσετε το Small Business Act για να στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης σας καλώ να προστατεύσετε τη βιομηχανία μας από την κινέζικη επίθεση. Πρέπει όμως να έχετε και νόμους κατά του dumping. Πρέπει να μπορούμε να αμυνθούμε έναντι των γιγάντων του διαδικτύου που πρέπει να πληρώνουν φόρους. Κατά τα άλλα, οφείλουμε να ενισχύσουμε και την γεωργική πολιτική πολιτική. Οι περικοπές στη γεωργική πολιτική είναι λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βιομηχανία και η γεωργία είναι δύο βασικά εργαλεία για να μπορούμε να έχουμε απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο ε, πρόσβαση στην πίστη. Οφείλουμε να έχουμε μία αγορά ε, των κεφαλαίων. Και όσον αφορά τη μετανάστευση, σα καλώ να σκεφτείτε αυτό το οποίο ψηφίστηκε επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο για την Αφρική. Το 2050 θα έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια Αφρικανούς. Αν δεν επέμβουμε σήμερα δεν θα βοηθάει ούτε η Frontex ούτε τίποτα άλλο. Ε, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τις ασθένειες, την τρομοκρατία. Αν η Ευρώπη λοιπόν δεν δραστηριοποιηθεί ε, θα έχουμε εδώ ροές δισεκατομμυρίων, όχι εκατομμυρίων ανθρώπων. Άρα πρέπει να κάνει πολλά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε περάσει 21, 21 μήνες από τη δολοφονία της δημοσιογράφου στη Μάλτα και ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι εντολή αυτή αυτής της δολοφονίας. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης ακόμα και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε τη Βενεζουέλα που έχουμε πολλούς Ιταλούς, Ισπανούς, Πορτογάλους και Γάλλους οι οποίοι εξακολουθούν να υποφέρουν λόγω τη δικτατορία στη χώρα. Και από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλει να ακούσει τη φωνή τους. Γιατί δεν είμαστε απλά μία ε, νοσή των αξιών. Είπατε κι εσεί τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν ακριβώ την κατεύθυνση. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Γκάια. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Φοντελάιν, ε, αναγκαστικά πρέπει να πω ότι στην επιστολή που μας στείλατε υιοθετείτε πάρα πολλά από τα αιτήματά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία αγωνιστήκαμε εμείς ως σοσιαλδημοκράτες και αυτά τα υιοθετήσατε. Μεταξύ άλλων, το επίδομα ανεργίας, ε, κάτι ε, το οποίο επιθυμεί διακαώς η δική σας πολιτική ομάδα. Αλλά αυτό επίσης υποκρύπτει το ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που αυτό το θέμα θέμα το υποτιμούν μέχρι να χαθεί τελείω. Και αυτό ισχύει κυρίω για χριστιανοδημοκρατικέ κυβερνήσει. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά που μα είπατε, εγώ τα αντιμετωπίζω επιφυλακτικά. Βεβαίω ε, θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχουν θεσμικά ουσιαστικά επιχειρήματα. Κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, εγώ στήριξα τον κύριο Τίμερμαν, τον Σπίτσεν Καντιντάτ και εκεί λοιπόν είχαμε κοινού στόχου, κοινέ αξίε. Ε, και εγώ εκεί δεν αποφάσισα με βάση την υπηκότητά μου. Υποσχέθηκα λοιπόν στους ε, ψηφοφόρου μου και αυτό το έκαναν όλοι οι υποψήφοι τη S5 ότι θα έχουμε και θα ψηφίσουμε μόνο έναν σπίτσαν καντιντάτ. Εμείς λοιπόν οι 16 προτιθέμεθα να τηρήσουμε αυτήν την υπόσχεσή μας. Πάρα πολλοί εδώ σε αυτό το χώρο επένεσαν το σπίτσαν καντιντάτ ως ε, ένα επίτευγμα της ε, Δημοκρατία. Σήμερα όμω είμαστε απογοητευμένοι και γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εσά Εσεί εσείς ε, πώς προτίθεστε να διασφαλίσετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί και δεν θα το επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει η κυρία Τσέχ. Thank you. It is a great... Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα που έρχομαι εδώ και είμαι εδώ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να κάνω όχι μόνο τα παρθενικά μου σχόλια αλλά τα, τα σχόλια του κόμματος μου στο Ρινιού. Είμαι ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία, μια πανέμορφη χώρα που δυστυχώς όμως ακούγεται για παραβιάσει του κράτου δικαίου ή τη δικαιμάδα Γενωνία των Πολιτών. Και φαντάζουμε πολλοί έχετε επιβδίσει. Το ίδιο και εγώ ως Ουγγαρέζα. Μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ελίτ εθελοτύφλησε αυτή η ευρωπαικη ελιτ εθελοτυφλησε απεναντι στον ε, λαϊκιστή Ορμπαν. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που προσπαθούν να καταστρέψουν την ένωσή μας και θα να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ένωση αξιών, να μείνουμε ενωμένοι, συσπηρωμένοι, ευήμεροι και ασφαλείς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ηγεσία που δεν θα φοβάται να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θέλουμε έργα και όχι μόνο λόγια. Η επόμενη επιτροπή θα πρέπει να δώσει τα εχέγγυα και τι ασφαλιστικέ δεκλίδε για να προασπίσει το κράτο δικαίου. Και οι ηγέτε, θέλουμε ηγέτε που θα έχουν την πολιτική βούληση να το εφαρμόσουν. Και Σήμερα μερικές φορές όταν κάθεται, ε, ε, φαίνεται κανείς στην Ευρώπη, ε, δεν λέει λόγια, αλλά δεν είναι αρκετά τα λόγια. Πρέπει να έχουμε πραγματική αλλαγή. Κυρία Βάνα. Κυρία Φαντελάη, είπατε πολλά για την ειρήνη στην Ευρώπη. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που ήταν, η ουδέτερη, την Αυστρία και ως πράσινη έναντι της ΠΕΣΚΟ και της Ευρωπαϊκής ε, Άμυνας και για τη συζήτηση για ένα στρατό και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ε, έναντι όλων αυτών είμαι ιδιαίτερα επικριτική και η πλειοψηφία των πολιτών της Ένωσης δεν θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα της Ένωσης η άμυνα. Θεωρεί ότι η εκπαίδευση, προστασία του κλίματος, τα κοινωνικά θέματα και πολλοί πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κυρίω να βασίζεται σε ανθρωπιστικά και διπλωματικά μέτρα για να αντιμετωπίζει τι ε, κρίσει στον κόσμο και όχι στρατιωτικά μέτρα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι λάθο να αυξάνονται συνεχώ οι δαπάνε τη Ένωση για αμυντικού σκοπού και για εξοπλισμού. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε επαρκεί ε, πόρου για την προστασία του κλίματος και για κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ εάν ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάβετε πρωτοβουλίες αφοπλισμού για να περιοριστούν οι αμυντικέ δαπάνες, ούτω ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα κοινωνικά και κλιματικά και για να υπάρχουν δεσμευτικοί έλεγχοι των εξαγωγών όπλων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Φάστ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Μινίστερ. Ευχαριστώ για την ομιλία σας νομίζω ότι θα έπρεπε να άνοιξε τα μάτια και των τελευταίων που δεν το πίστευαν ότι είστε το λάθος άτομο για αυτή τη θέση. Και το ΕΛΚ μοιάζει να έχει γίνει τώρα μια πράσινη ομάδα. Το κείμενο το οποίο μας στείλατε είναι πραγματικά μνημείο οπορτουνισμού. Όλα θα γίνουν σωστά, ισότητα φίλων βιώσιμη Ευρώπη ένα κοινοβούλιο των παιδιών, μη του, θα ενισχύσετε τις μεσαίες τάξεις. Όλα αυτά μοιάζει να είναι οι κοινοτοπίες ε, των πράσινων και αριστερών. Και το πρόβλημα είστε και εσείς, οι θέση σας. Αυτή η εντύπωση δίνεται ότι προσπαθείτε να τα επιτύχετε όλα και τίποτα. Και η ταυτότητα της Ευρώπης, η ταυτότητα ως πατρίδα χάνονται όλα αυτά σας ενδιαφέρει μόνο να πάρετε μια καινούργια θέση, ένα νέο πολιτικό τρόπεο και ένα νέο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Τι θέλετε λοιπόν εδώ μέσα. Με την ομιλία που κάνατε πρέπει όλοι να είστε προετοιμασμένοι, ε, να, έχετε πάρει όλο το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατόν να κλέξετε αυτή τη γυναίκα ως πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο κύριο Τέρτς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντελάιεν, Όλοι είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι και ανησυχούμε γιατί βλέπουμε ότι στην ουσία δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του κυρίου μας και της ε, κυρίας Βαντερλάιεν, των δύο υποψηφίων. Γιατί προσπαθήσατε σήμερα με την ομιλία σας ε, να ικανοποιήσετε την αριστερά πτέρυγα, τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές και μάλιστα τους στείλατε επιστολή με εξηγήσει για το σχέδιό σας. Αλλά προς την άλλη πτέρυγα δεν στραφήκατε. Και Εκεί έχουμε πραγματικά σοβαρή κατάσταση. Ήδη, κυρία Βαντελάιεν, εφαρμόσατε αυτό τον υγειονομικό κλειό, αυτόν τον αποκλεισμό ενός τμήματος των Ευρωπαίων με τη συμπεριφορά σας. Γιατί διαπιστώνουμε ότι ε, ε, υιοθετείται μια συμπεριφορά που τιμωρεί τους λαούς που εκλέγουν κυβερνήσεις που δεν είναι της αρεσκίας κάποιων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ επικίνδυνο και βλέπουμε πώς ε, τιμωρείται κάποια κόμματα που έχουν εκλεγεί από το λαό με πολιτική και απόψεις που δεν είναι της αρεσκίας κάποιων δεν είναι της αρεσκίας της πλειοψηφίας που δημιουργήθηκε εδώ σε αυτή τη συνένεση όπου ο Τίμερμαν μας και εσείς είστε το ίδιο ακριβώ. είστε το ίδιο ακριβώ και το Μόνο ο στόχος είναι να περιθωριοποιήσετε κάποιο, κάποιους άλλους. Και ουσιαστικά βρίσκεστε απέναντι, είπατε, σε εκείνους που είναι κατά της ε, ενότητας. Ε, νομίζω ότι ε, το χειρότερο πλήγμα στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χειρότερο πλήγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό ο υγειονομικός κλειός, αυτός ο αποκλεισμό που εφαρμόζεται, που δυναμητίζουν το δημοκρατικό πνεύμα, δυναμητίζουν τους κανόνες και σε τελική ανάλυση δια, ε, δυναμητίζουν οποιαδήποτε ενθουσιασμό και όραμα για ένα κοινό σχέδιο. Ο κύριος ε, Γιώργη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από εμά ε, θεώρησαν το Brexit ένα δίδαγμα και μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ. Ένα σήμα ότι χρειάζεται επιγόντως αλλαγή πορείας. Πολύ εύλογα είναι δυσαρεστημένοι οι Ευρωπαίοι πολίτε από την αδιαφανή και αντιδημοκρατική λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα. Κυρία Βαντελάιεν, είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε το σύστημα των σπίτσεν candidate των κορυφαίων υποψηφίων. Αυτό ήταν τραγική ηρωνία, για να μην πω ότι ήταν και κοινικότητα. Γιατί αυτό το σύστημα ουσιαστικά παραβιάστηκε για να διοριστείτε εσεί υποψήφια. Το σύστημα του σπίτσεν candidate των κορυφαίων υποψηφίων μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση για την επιλογή ενό υποψηφίου για την ε, Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική σα υποψηφιότητα δείχνει ότι ηγέτε ε, των Ευρωπαϊκών κρατών αγνόησαν το εκλογικό σώμα και δεν έμαθαν από τα προηγούμενά τους παθήματα. Γιατί τέτοια λάθη δείχνουν άγνοια και κοφεύουν απέναντι στον ευρωσκεπτικισμό. Ε, οπότε ε, Επίσης απογοητεύσατε αυτούς που θέλουν μια ισχυρότερη, πιο αξιόπιστη, πιο δημοκρατική και διαφανέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βαντερ Λάιεν, δεν φταίτε εσείς βέβαια. Αλλά συμβάλλατε σίγουρα τα μάλα σε αυτή την απογοήτευση. Και γι' αυτό πολλοί ευρωβουλευτές ε, κρίνουν απαράδεκτη την υποψηφιότητά σας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριο Σρανζέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βαντερ Λάιεν για την ε, ομιλία της που μας ενέπνευσε, ήταν πολύ και εμπνευσμένη και έδειξε πραγματικά ευρωπαϊκή δέσμευση και αφοσίωση. Και σα διαβεβαιώ ότι θα έχετε την υποστήριξή μα. Έχω όμω δύο παρατηρήσει. Καταρχήν, λυπάμαι που ενώ είστε ε, γιατρό και έχετε ιδιαίτερε ευαισθησίε για την υγεία, δεν κάνατε ούτε την παραμικρή μνήμα στο master plan που ε, υπέβαλε στην προεκλογή του εξαιρετία το ΕΛΚ για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτή ήταν σημαντική φιλοδοξία του κόμματό μα και ελπίζουμε να το αισθενιστεί και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτου λεχθέντο έχω και μία ερώτηση που για μένα έχει θεμελιώδη σημασία. Ε, γιατί δεν απαντήθηκε από κανέναν. Ε, ε, μιλήσατε για το σεβασμό του ΠΔΠ, τι δημοσιονομικέ προοπτικέ για την περίοδο 2021-2027. Στην ουσία όμως αυτό που διαπιστώνουμε στις στην πολιτική της συνοχή είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άδικη. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, μια χώρα όπως η Ιταλία ε, που είναι στη μέση ώρα έχει το 6% ε, της συνοχής, η Κροατία 16%. Η Φιλανδία που είναι πολύ πάνω από το κοινοτικό μέσο όρο λαμβάνει 5% της πολιτικής συνοχής. Μια χώρα σαν τη Λιθουανία 23%. Και μιλώ για γειτονικέ χώρες που μπορούμε να τις συγκρίνουμε για να ε, διαπιστώσετε ότι είναι άδικη η πολιτική συνοχής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, γιατί 45% ε, του Ευρωπαϊκού Κονδυλίου της Συνοχής το άφησε χωρίς εξηγήσει. Και επίσης ε, για την ε, συγχώνευση του ΦΕΝΤΕΡ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δημιουργούνται πολλά προβλήματα κοινωνικά και για την πολιτική συνοχή. Κυρία Βανταράιν, το θέμα τη συνοχή και τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών έχει θεμελιώδη σημασία, γιατί απευθύνεται μια έκκληση για την ενότητα. Αν όμω δεν αναθεωρηθούν οι δημοσιονομικέ προοπτικέ προ την κατεύθυνση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σα διαβεβαιώ ότι θα υπάρξουν και προβλήματα συνοχή και προβλήματα ενότητα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Σα ευχαριστώ. Madame Guillaume, one minute. Η κυρία Κιγιόμ για ένα λεπτό. Κυρία Βαρτενλάγερ, κάνετε μία αρκετά άρτια παρουσίαση. Ε, συμπληρώστε αρκετά κουτιά, αλλά όχι όλα. Διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Και είστε εδώ διότι ξεκίνησε μια διαδικασία ε, υποψηφιότητά σας αρκετά ιδιόρυθμη Υπάρχουν ε, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι παρόντε εδώ για να σα υποστηρίξουν, ε, που είναι αυτοί οι οποίοι σα υποστήριξαν. Το Συμβούλιο δεν έλαβε καθόλου υπόψη την ε, γνώμη των πολιτών, οι οποίοι ψήφισαν το speech and candidate για να του εκπροσωπήσει. Και ουσιαστικά υποβαθμίζεται και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πλέον ένα junior partner στην όλη επιχείρηση. Όσον αφορά τα θέματα μετανάστευση και ασύλου, δεν αρκεί να μα λέτε ότι θέλετε να μεταρρυθμίσετε για νιωστή φορά το πακέτο για το άσυλο, το οποίο μεταρρυθμίστηκε και ξαναμεταρρυθμίστηκε και πλέον δεν καταλαβαίνει κανεί τι λέει. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση διάθρωση στη θάλασσα, η οποία θα σώσει και την αξιοπρέπεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον και του Συμβουλίου. Ε, αυτό θα δείξει ότι είστε διατεθειμένοι να δώσετε τη μάχη και να αλλάξετε και το πρόσωπο τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέντερ λέει για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Βαντερ Λάιεν, πρέπει να πω κάποια πράγματα ειλικρινώ. Εγώ ήμουν αρκετά επικριτικό ε, στην υποψηφιότητά σα. Ε, ήμουν αρκετά επικριτικό ε, και στο γεγονό ότι θα γίνεται ίσω επικεφαλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η διαδικασία αυτή με έκανε να νιώσω ότι υπάρχει σεβασμό στη θέση μου ω Ευρωβουλευτή και ω εκπρόσωπο των Σουηδών ψηφοφόρων. Γι' αυτό σα επενώ. Αλλά υπάρχει και μία νέα ομάδα η οποία θέλει να ε, νικήσει τους λαϊκιστές ε, σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς και θα λάβετε την ψήφο μου σήμερα, διότι φαίνεται να δείχνετε ειλικρινό ενδιαφέρον για το τι πιστεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θυμάμαι και τη διαδικασία πριν από πέντε χρόνια. Δεν νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι ένιωσαν ότι υπήρχε ε, κατάλληλο διάλογο με τον υποψήφιο πρόεδρο τη τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Γιούνκερ. Ενώ είναι σωστό ο διάλογο μαζί σα και γι' αυτό σα σέβομαι. θα πρέπει όμω να λάβετε και κάποιε πρωτοβουλίε. Για παράδειγμα, έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να υπάρχει νομοθεσία για την ευημερία των ζώων εδώ και πέντε χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα από αυτού μέχρι τούδε. Επομένω, θα επανέλθουμε μόλι θα συσταθεί το Σώμα των Επιτρόπων και θα επαναλάβουμε το αίτημά μα και θα είστε και υπόλογοι από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σκοτκάτο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτοί που θέλουν να σταματήσουν την ε, καταστροφική έξοδο της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για αυτό που ακούσατε. χάρηκα που είπατε ότι θέλετε να μας δώσετε τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται και είστε υπέρ της παραμονής μας για να διασώσουμε αυτή την ε, ζωφερή στιγμή στην ιστορία της χώρας μας. Όσον αφορά την προστασία της ζωή ε, τη χλωρίδα και τη πανίδα. υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτό που πρεσβεύετε εσεί και που πρεσβεύουν οι πράσινοι. Δυστυχώ, εγώ δεν θα μπορώ να σα υπερψηφίσω. Αυτή η συμφωνία η οποία έγινε στο περιθώριο ε, και κρυφά ε, στο Συμβούλιο δεν βοηθάει διότι απειλείται το κράτο δικαίου και οι δημοκρατικέ αξίε. Είναι λυπηρό το γεγονό ότι θα εξαρτώνται από την ψήφο τη ακροδεξιά και όχι τη ισχυρή φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία που θα μπορούσε μπορούσαμε να έχουμε αν έχετε την ριζοσπαστική αλλαγή που ζητούν οι πράσινοι ψηφοφόροι. Για ένα λεπτό, Άντερσον. Η κυρία Άντερσον. Να, δεν είναι εδώ. Α, καλημέρα σας. Κυρία ε, Υπουργέ, θα είμαι σύντομη. Είστε λάθος πρόταση από κάθε άποψη για οποιοδήποτε αξίωμα. Έχετε αναλάβει διάφορες άχρηστες πρωτοβουλίες και δαπανίσατε δημόσια χρήματα για να χρηματοδοτήσετε διαφημιστικές εταιρείες για να ασκήσουν πίεση στην ε, γερμανική κοινή γνώμη. Οι στρατιώτες σας ε, δεν έχουν καθόλου ηθικό. Έχετε ευνουχίσει τον γερμανικό στρατό. Και φροντίσατε να υπάρχουν διάφορες δυνατότητες βρεφονιπιακών σταθμών. Μετατρέψατε τον γερμανικό στρατό σε ένα γελίο βρεφονιπιακό στρατό. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ε, θέλει να εκλεγείται. Δεν θέλω λοιπόν να εκλεγείτε για να μην συνεχίσετε το καταστροφικό σας έργο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να βασιστείτε στη δική μου στήριξη. Παρακαλώ να το σημειώσετε. Εγώ εγώ είμαι πεπισμένη ότι δεν είναι δυνατόν να σας ψηφίσω. Θα προτιμούσα να μου κόψουν το χέρι. Ήμουν για πολύ καιρό ψηφοφόρος του Τσεντεού, όχι πια. Ευχαριστώ πολύ. Βαν Όρντεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρα Φοντερ Λάιν, με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που είπατε ότι θέλετε να υπάρξει ευρωπαϊκό στρατό και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αυτό είναι ένα πολιτικό εγχείρημα θα οδηγήσει σε διχασμό μεταξύ τη Ευρώπη και των ε, βόρειοαμερικανών αμερικανων συμμάχων μας και θα υπονομεύσει τον ΝΑΤΟ. Αλλά κάποια κρίσιμα θέματα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλωσορίζουμε τη δήλωσή σα ότι σέβεστε την απόφαση του Βρετανικού λαού να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανάγκη ότι πρέπει να συνεργαστείτε στενά με την Βρετανία στο μέλλον, γιατί η καλή θέληση από πλευρά Βρυξελών ε, δεν υπήρξε μέχρι τώρα. Αλλά λυπόμαστε που το μόνο που, πρέπει να, που βλέπουμε να προτείνεται είναι να παραταθεί η προθεσμία αποχώρηση. Δεν είναι πολύ φιλόδοξο αυτό. Θα ήθελα παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σα, ώστε να υπάρξει αναθεώρηση ή επανερμηνία των ε, σημείων τη συμφωνία αποχώρηση που είναι καθαρά απαράδεκτα Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θέλει πολύ χρόνο αυτό. Υπάρχουν λύσει. Στην Ευρώπη, όπω λέγεται, τίποτα δεν είναι δυνατόν και όλα δυνατά. Η Βρετανία θα αποχωρήσει στι 31 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α διασφαλίσουμε ότι θα γίνει με καλού όρου, χωρί αντιδικία, για να υπάρξει μια βάση για μια ε, ισχυρή θετική σχέση στο παρελθόν. Με πλήρη σεβασμό προ την βούληση του Βρετανικού λαού για τον έλεγχο των νόμων και των συνόρων του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κόλα Κούσιτ. Σα ευχαριστώ το θεμέλιο ε, της ανάπτυξης ε, και της πρόοδου αλλά και της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενότητα και το κράτος δικαίου. Η ενότητα και το κράτος δικαίου ε, φυσικά φαίνονται από τον τρόπο και αντικατοπτρίζονται στον τρόπο εκλογής του Προέδρου από τους τις τέσσερις βασικές ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι τρεις ε, πέρασαν στη Γερμανία. Στην Σλοβακία και την Κροατία τίποτα, μηδέν. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να δοθούν θέσεις με βάση και τη γεωγραφική εξισορρόπηση. Οπότε έχει εδώ παραβιαστεί και θυγεί και το κράτος δικαίου. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Έχουμε τη Γερμανία που έχει 20 εκπροσώπους εκπροσώπους. Ε, κάτι που είναι αντίθετο με την ενότητα, γιατί δημιουργεί υπεροχή. Και επιπλέον θέλουμε να εκλέξουμε και πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γεωργία. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο, γιατί δεν αντικατοπτρίζει την Ευρώπη της ενότητας. Και δυστυχώ μια τέτοια Ευρώπη θέτει αναφιβόλω την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, κυρία Δελάγκη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εκλογές στην Ολλανδία α, μας έδειξαν γρήγορα ότι αν θέλει κανείς να παραμείνει στο πόστο του θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Ακούσατε κυρία Φόντερ Λάινεν, κάποιους να λένε ότι τα σχέδιά σας παρά είναι φιλόδοξα και άλλους να λένε ότι υπολείπονται του ζητούμενου. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια σωστή ισορροπία Πολλά μας είπατε στην παρουσίασή σας για τις προτάσεις σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει και την αυτοκριτική του. Η υποψήφιος μίλησε για την αξία της ενότητας και αυτή την ενότητα δεν την διαπιστώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι ο Σπίτσεν το κορυφαίο υποψήφιο του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος, μπορεί να προωθεί ή τουλάχιστον να περάσει ο δεύτερος ε, Spitzenkandidat. Είναι όμω αφελές να πιστεύουμε κάτι τέτοιο, γιατί ε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη διαφάνεια το ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μερικοί απλώ προβάλλουν ε, τη δική τους θέση. Μακρόν και Ορμπάν, πολύ περίεργο και αλόκοτο συνδυασμό. Και όμω αυτοί ουσιαστικά επικράτησαν. Ακούσαμε από την υποψήφιο ότι θέλει να διορθώσει τη ζημιά που έκανε το Συμβούλιο και να την περιορίσει ε, για το 2024. Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας, ε, ε, μιλήσατε για τη Σιμών Βάιλ, που δεν ήταν μόνο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και από τις πρώτες ελάχιστες δυστυχώς γυναίκες της, μέλη της Γαλλικής Ακαδημίας. Και όταν έγινε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας έλαβε ένα σπαθί και στο σπαθί φρόντισε να χαράξει τρία πράγματα. 7, 8, 5, 6, 1. Τον αριθμό της δηλαδή στο Auschwitz. Και να θυμάται ε, να θυμόμαστε κάθε μέρα γιατί έχουμε την Ευρώπη και γιατί θα πρέπει να δίνουμε καθημερινά μάχη για αυτή. Το σύνθημα της γαλλικής δημοκρατίας και το σύνθημα της Ευρώπης είναι η ενότητα στην πολυμορφία. Και η επιλογή που έχουμε να κάνουμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, το βράδυ, ε, για όσου από εμά είμαστε υπεύθυνοι και επικοδομητικοί είναι θα καθοδηγηθούμε στην, στην ψήφο μας από την απογοήτευση, τη ματέωση και τον θυμό για την εκρυπτό και παραβίστο συμφωνία του Συμβουλίου ή θα διαπνόμαστε από το πνεύμα της Σιμών Βαέλ ε, και που θέλει αυτή η υποψήφιος ε, να πραγματώσει δηλαδή την Ευρώπη που, που χρειάζονται οι πολίτες. Ευχαριστώ κυρία Μποναφέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, συνάδελφοι, να σας πάω λίγο πίσω στις ευρωεκλογέ το Μάιο, όταν τα εθνικιστικά κόμματα τα οποία υπέβαλαν ε, ψηφιότητα, οι οποίοι έδιναν στίχημα για την αποτυχία και την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επέτυχαν το σκοπό του τουλάχιστον προς το παρόν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να πιστέψουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς, κυρία Βοντερ ζητάμε να σταθείτε στο ύψος ε, αυτού του στόχου, να δώσετε μια ισχυρή ένδειξη τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πέραν του γεγονότος ότι για πρώτη φορά μια γυναίκα θα είναι πρόεδρος ενός τόσο πολύ σημαντικού θεσμικού οργάνου. Και να σα το πω με δύο λόγια. Θέλουμε μια ευρωστή και λέγε Ευρώπη, η οποία δεν θα γυρίζει πλέον ε, ε, στην άλλη πλευρά για όσου μένουν πίσω, αλλά θα έχει το σθένος να χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για να υπάρξει επιτέλου ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη, το οποίο χωρί αμφιβολία θα θέσει και τα περιβαλλοντικά θέματα. Όχι περιθωριακά όπω βλέπουμε πολλέ φορέ και εδώ, αλλά ω ευκαιρία ε, που δεν ανακόπτει αλλά αυξάνει την ανάπτυξη γιατί την κάνει βιώσιμη. Και έτσι εσείς ε, θα μπορέσετε να απαντήσετε και σε όλους εκείνους που είπαν ακόμα και εδώ σήμερα ότι υπεκφεύγετε. Ε, θέλουμε λοιπόν να μην ε, ε χάσετε από τους εθνικιστές, ε, να κρατήσετε σταθερή την σημαία του ευρωπαϊσμού η οποία γίνεται από ευθύνε. και όταν μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση αλλά και όταν μιλάμε και για τη μετανάστευση. Το κάναμε εδώ στο Κοινοβούλιο όταν ζητήσαμε τροποποίηση του συστήματος του Διβλίνου. Μόνο ε, αν αυτό είναι το όραμα και η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας στηρίξουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Χανσάροβα για ένα λεπτό. Χαράνσοβα, συγγνώμη. Κυρία Υποψήφια Πρόεδρε, πριν από 15 χρόνια ε, οι κεντροευρωπαίοι έδωσαν εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τώρα αυτή η εμπιστοσύνη αρχίζει να διαβρώνεται. Ε, πολλά πράγματα στο παρελθόν δημιούργησαν ένα χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ε, για διάφορους λόγους. Ενιαία αγορά, διπλή ποιότητα των προϊόντων, απόσπαση των εργαζομένων, όλα τα θέματα της πιο ασφαλούς Ευρώπης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια νέα ε, ε, διαφορετική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορέσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη που έχουν χάσει οι πολίτες, να εξασφαλίσει ότι τίνουμε βίκονους ε, σε ό,τι έχει να πει ο καθένας πριν γίνει οποιαδήποτε πρόταση και να συνεχίσουμε να καταργούμε τα υφιστόμενα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και όχι να δημιουργούμε νέα προσκόμματα. Να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες με τον ίδιο τρόπο να έχουν ίση πρόσβαση σε εργασία και σπουδές οπουδήποτε στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν, ε, κύριε υποψήφια πρόεδρε, ελπίζω να μπορέσετε σήμερα να γίνετε η φωνή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρτασούν για ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, πολύ καλημέρα σας. Η υποψηφιότητά σας είναι μια τριπλή ε, εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη της ε, κοινοβουλευτικοποίησης της δημόσιας ζωής και εγκατάλειψη του ισχυρού κράτους δικαίου. <clears throat> Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο κύριος Τίμερμανς δεν είναι εδώ ε, επειδή κάποια κράτη-μέλη πρότειναν βέτο επειδή ήθελε να επικρατήσει το κράτος δικαίου. Επιπλέον η Επιτροπή θα ξεκινήσει με ένα αρχικό ατόπιμα αν εκλεγεί με κάποιες ψήφους από την ακροδεξιά. Γιατί κάτι τέτοιο θα αμφισβητήσει τον αποκλεισμό της ακροδεξιάς που προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε αυτό το σώμα. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν μπορώ να σας ψηφίσω. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να την απορρίψει. Και σε όσους μας λένε ότι για λόγους φιλοευρωπαϊσμού πρέπει να σας στηρίξουμε, πρέπει να σας πω ότι πάντα να υποβάλλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επιπτώσεις ε, των κακών αποφάσεων του Συμβουλίου είναι η χειρότερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στην Ευρώπη. Για λόγους ε, στήριξης της Ευρώπης και των θεσμών και των διαδικασιών θα πρέπει το Συμβούλιο να μας κάνει μια νέα πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρά. Ένα λεπτό. Κυρία υποψηφία, κυρίες και κύριοι, τι βλέπουμε εδώ. Είναι, είναι πραγματικά υπόδειγμα του τι δεν πρέπει να κάνουμε. τι υποσχέσεις μας δόθηκαν για δημοκρατία μέσω του συστήματος ε, Candidate. Αν εκλέξουμε την κυρία Φόντερ Λάιεν, στην ουσία τα απορρίπτουμε όλα αυτά. Είναι ένα παιχνίδι. Κύριε Βέμπερ, εσείς ε, είπατε ότι θα είστε speech and Candidate. Και τώρα συγχαίρετε την κυρία Φόντερ Λάιεν και τη λέτε ότι θα τη στηρίξετε. Δηλαδή, τι αξιοπρέπεια είναι αυτή. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την καριέρα της κυρίας Φόντερ Λάιν ξέρουν ότι ο Υπουργό Άμυνας απέτυχε πλήρως. Ο γερμανικός στρατός έχει τώρα αεροπλάνα που δεν πετάνε, όπλα που δεν πυροβολούν, τάγκ που δεν μπορούν να κουνηθούν. Τι να πω. Σε αυτούς που θα σας ψηφίσουν να πω μόνο ένα πράγμα μεγαλύτερο, ε, η μεγαλύτερη υπονόμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μπορούσατε να κάνετε παρά να εκλέξετε μίαν που απέτυχε ως Υπουργός στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιεν, Μα παρουσιάσετε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, αλλά ελάχιστα μα είπατε για το πώ σκοπεύετε να το εφαρμόσετε. Για κάποιε στιγμέ με επαναφέρατε στην παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα στη σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία και εκεί είχα πολλέ ευκαιρίε να ακούσω κάποιε υψηπετεί ιδέε παρόμοιε με τι δικέ σα. Αδελφότητα και ενότητα, πολιτική ολοκλήρωση, κοινό στρατό, περισσότερα δικαιώματα για του εργαζόμενου και τι γυναίκε και γνωρίζουμε τι κατάληξη είχαν όλα αυτά. Έτσι θα, εκεί θα καταλήξει και το δικό σας όραμα, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Αν το ήθελαν, δεν θα φοβόσασταν σήμερα αν θα συγκεντρώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλειοψηφία. Μιλάτε για την ενότητα και την ισότητα στην Ευρώπη και ξεχνάτε ότι όλες τις ηγετικέ θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελέχωσαν ε, μέλη από τις παλιότερες χώρες μέλη. Αυτά για την ενότητα. Και θέλετε αλλαγή τη τρόπου ψηφοφορία στην εξωτερική πολιτική. Αυτά για την ενότητα. Επίσης αναφέρετε τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκής, ε, της της Ευρώπη, την ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Αλλά ως χριστιανοδημοκράτησα, ξεχάσατε το χριστιανισμό. Φαίνεται ότι η Ευρώπη σα φεύγει μακριά και απομακρύνεται από τις καταβολές της. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένη στη διάλυση. Ευχαριστώ κύριο Τζαρούσο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Κυρία Βαντελάιεν, μας ζητάτε εμπιστοσύνη, αλλά η εμπιστοσύνη μα δεν θα γίνει ποτέ εν κρυπτό, ούτε θα είναι δεδομένη, ούτε για ένα λεπτό. Θα αποτελέσει όπλο για να μπορέσουμε να ε, ελέγχουμε την πολιτική σα. Ακούσαμε για μια δίκαιη πολιτική, ακούσαμε για Ευρώπη των εργαζομένων και του περιβάλλοντο. Λέτε ότι θα σώσετε και ανθρώπινε ζωέ και θα μεταρρυθμίσετε τη μετανάστευση και το άσυλο. Ναι, πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και δεν μπορούμε πλέον σε μια χώρα να ρίχνουμε το βάρο τη μετανάστευση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει αυτό που ε, έγινε ε, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει γίνει αυτό. Ε, η ανεργία των νέων στην Ιταλία είναι πολύ ψηλή και δύσκολα ένα νέο μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Κυρία Βαντελάιν, θέλουμε επιτέλου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει σε όλου του γεωργού, του αλληλεί, του εργαζομένου, του νέου, σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε όλε τι ευκαιρίε ανάπτυξη. Γι' αυτό θα σα ζητήσουμε μια σοβαρή και συγκεκριμένη δέσμευση για να σταματήσουν η φορολογική παράδοση, για εναρμόνιση των πολιτικών ε, τη φορολογία και ε, μια πολιτική κατά τη μαφία πολύ αυστηρή. Αν πολλά από αυτά τα οποία Μα είπατε στην αρχική σας παρέμβαση, μπορείτε πραγματικά να βασίζεστε στη στήριξή μας. Αλλά εάν παραμείνουν κενά γράμμα και απλώς τιμωρείτε την Ευρώπη όπως τιμωρήσατε και την Νότια Ιταλία, το, το κίνημα των πέντε αστέρων πραγματικά θα είναι η πιο ισχυρή σας αντιπολίτευση. Ο κύριος Τομπέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Βοντελαέν. Πραγματικά ελπίζω όλοι σήμερα που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία, πιστεύω ότι όλοι θα σας δώσουν τη στήριξή τους σήμερα η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά φαίνεται ότι θα σας καταψηφίσουν σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το θεωρήσετε ως ε, τίτλο τιμής για σας. Ε, σας τιμά κατά κάποιο τρόπο. Από ό,τι φαίνεται οι πράσινοι όμως ε, στρατεύονται με αυτούς και πραγματικά με εκπλήσει αυτό και πρέπει να πω ότι ντρέπομαι και λίγο διότι θα καταψηφίσετε την πρώτη γυναίκα υποψήφια πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, επειδή κάποιο ο οποίος θα μπορέσει να έχει μια πλειοψηφία για μια κλιματική πολιτική για την Ευρώπη είστε εσεί. Ε, πραγματικά λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε στην Ευρώπη και το κλίμα αλλά και το διασυνοριακό έγκλημα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, και θέματα που πλήττουν την ελευθερία ε, μετακίνηση. Ε, δεν θα πρέπει φυσικά η ελεύθερη ε, κυκλοφορία ανθρώπων να είναι και ε, κάτι το οποίο θα βοηθά το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να αποτελούν ουσιαστικό θέμα όλα αυτά Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλε πλειοψηφίε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ταυτόχρονα και καλύτερο έλεγχο για την μεταναστευτική πολιτική μα. Είμαι βέβαιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να έχει την κατάλληλη πλειοψηφία για να υποστηρίξει μια μεταναστευτική πολιτική η οποία θα γίνεται και με την καρδιά και με το μυαλό. Τέλο, επιτρέψτε μου να πω ότι η Ευρώπη για μένα αφορά την ελευθερία, αφορά την επιχειρηματικότητα, ε, το γεγονό ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και προστασία για όλους μας τους πολίτες. Θα έχετε λοιπόν την υποστήριξή μας κυρία μου σήμερα και βέβαια ε, πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πρέπει να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Καλιοράντ, για ένα λεπτό. Κυρία Φοντερ Λάιεν, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις που κάνατε σήμερα και για την επιστολή που στείλατε στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έτυχε ε, καλής υποδοχής και συνέβαλε ε, τα μάλα στην συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στι Βρυξέλλε. Αναγνωρίζω τη δέσμευσή σα υπέρ τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, μια δίκαιη και ισότιμη Ευρώπη, χωρί διαχωριστικέ γραμμέ. Και τώρα πραγματικά ε, αδειμονώ για συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοί μου. Επίσης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε, μια άλλη διαχωριστική γραμμή που δεν αναφέρατε σήμερα στην ομιλία σας. Της ε, διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ε, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου όλες οι σημαντικές θέσεις, οι θύνουσες θέσεις, δόθηκαν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δεν θέλουμε μία Ευρώπη που χωρίζεται σε Ανατολή και Δύση ή σε χώρες με περισσότερες ψήφους και λιγότερες ψήφους. Δεν μπορούμε έτσι να χτίσουμε την Ευρώπη. Γι' αυτό και σας ε, ερωτώ πώς ε, αξιολογείτε εσείς αυτή την απόφαση και τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποφύγουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή και να μην την ευαθύνουμε κιόλας. Ο κύριος Γκινέα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιεν. Έκλεισε το μικρόφωνο δυστυχώς. Μάλιστα. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι πολύ σημαντικό για τη ρουμανική αντιπροσωπεία. Το θέμα της ε, οικονομικής και ε, δημοσιονομικής ολοκλήρωσης. Ε, το Προπολογισμό της Ευρωζώνης και χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη, όπως η Ρουμανία. Χρειαζόμαστε κάποια υποστήριξη ε, και κάποια τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να ενταχθούμε απρόσκοπτα στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Γιούγκερ αναφέρθηκε επανειλημμένος ε, σε αυτό. Χαιρετίζω την πρόθεσή σας ε, να προτείνεται ένα πανευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο και για τη δική μας ομάδα, το Renew Europe, την ε, ανανέωση της Ευρώπης. Και μάλιστα είχαμε προτείνει αυτό το μηχανισμό πριν από δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα χρειαζόμασταν τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Σμιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουν όλα υποθεί, αλλά δεν έχουν όλα υποθεί από όλους. Κυρία Φόντερ Λάιν, να σας συγχαρώ. Εντυπωσιακή η ομιλία σας σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι έχετε προχωρήσει πολύ στην ε, συζήτηση με τις ομάδες. Ιδιαίτερα η δέσμευσή σας για ένα σώμα επιτρόπων με ίσο αριθμό ανθρώπων και γυναικών. Αυτό ε, θα είναι σημαντική αλλαγή. Η σκοτσέζικη κυβέρνηση είχε εδώ και πέντε χρόνια ίσο αριθμό ανδρών γυναικών. Θετικό. Για τον Brexit θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι συνάδελφοι στην Αγγλία, στην ε, Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και αλλού προσπαθούν να κάνουν αυτούς που είναι υπέρ του Brexit να δουν λίγο λογική. Το καλύτερο Brexit είναι όχι Brexit. Ορισμένοι προσπαθούμε να βρούμε πραγματικές λύσεις και χαίρομαι που θα είστε σύμμαχος ε, κρατώντας την πόρτα ανοιχτή για μας. Ε, κάτι άλλο. Δεν είναι το σώμα μας πλήρες. Δεν έχουμε τρει συναδέλφου από την Καταλωνία, τον συνάδελφο Γιουνκέρα για παράδειγμα. Η μόνη λύση για αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα είναι ο διάλογο. Και εσεί προσωπικά είστε σε θέση να παίξετε το ρόλο εντύμου διαμεσολαβητή και ελπίζω να τον παίξετε σε αυτόν τον διάλογο. Ευχαριστώ πολύ.